El señor Αγαπητές φίλες και φίλοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ξεκινήσουμε τι συνεδρίες. Το πρώτο σημείο είναι η έκθεση Γκέριγκερ Ντεότεμπεργκ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκέριγκερ. Έχει έξι λεπτά η κυρία Γκέριγκερ Ντεότενμπεργκ στη διάθεσή της, τέσσερα λεπτά στην πρώτη φάση και δύο λεπτά εκ των υστέρων. Αυτό είναι μια σύσταση βέβαια, να μιλήσετε τέσσερα λεπτά στην πρωτολογία σας και μετά να ακολουθήσουν άλλα δύο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο πλαίσιο της ε, επικουρικότητας ε, θα πρέπει βεβαίω να βελτιώσουμε την νομοθεσία, θα πρέπει η νομοθεσία να είναι σαφής, ξεκάθαρη και κατανοητή, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Το ευρωπαϊκό δίκαιο συχνά περιγράφεται ως μη ακριβές και με περιπλοκές και λένε συχνά πως ε, αφήνει πάρα πολύ μεγάλα περιθώρια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του άρθρου 260 στην ε, συνθήκη, σύμφωνα με το οποίο μπορεί η Κομισιόν ε, να επιβλέπει την εφαρμογή και να κάνει αναλογέ συστάσει στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό χαιρόμαστε για αυτά τα οποία είπε και για τον κανονισμό που έφερε πέρσι ο κύριος Μπαρόζο. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την ε, Κομισιόν τι κάνει συγκεκριμένα. Το θέμα αυτό δεν ε, ελπίζω να μην ήταν μόνο τυπικότητες. Το επόμενο θέμα το οποίο πρότεινε ο κύριος Μπαρόζο ήταν μια αξιολόγηση ex post και πράγματι πρέπει να δούμε τι γίνεται και μετά την έγκριση της νομοθεσίας, αν εφαρμόζεται αυτή σωστά και τι προκύπτει και από πού ε, προέρχονται οι καθυστερήσεις, εάν ε, δεν ε, επιδρά σωστά στην κοινωνία, στην οικονομία, στο περιβάλλον, τότε η δουλειά μας δεν έχει κανένα νόημα. Το επόμενο λοιπόν ερώτημά μου προς την Κομισιόν είναι τι γίνεται με την αξιολόγηση εξπόστη και ποια είναι η διαφορά με την αξιολόγηση που γινόταν μέχρι τώρα. Ε, προσέχει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα να γίνεται η σωστή αξιολόγηση αντικτύπου από την ε, Κομισιόν και αυτό πάντα εγώ το έβλεπα υποδιοπτυχές πρώτα απ' όλα από την πλευρά της ουσίας. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση όντω των αντικτύπων, ειδικά όσον αφορά τον κοινωνικό αντίκτυπο και Σημαντική βεβαίως είναι η απάντηση εδώ πέρα στο τι γίνεται στις διάφορες αγορές εργασίες και στους διάφορους τομείς αγοράς εργασίες, ειδικά υπό την πτυχή της οικονομικής κρίσης. Νομίζω πως δεν έχει ερευνηθεί αρκετά αυτή η πτυχή και η άλλη πτυχή είναι η ανεξαρτησία των αξιολόγιων αυτών γιατί θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης ανεξαρτησία. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τους πόρους που θα πρέπει να δίνονται για αυτή την αποστολή. Ο Πρόεδρος, οι διερμηνείς μου λένε πώς μιλάτε λίγο γρήγορα. Ε, θα προσπαθήσω κύριε Πρόεδρε, αλλά ε, είχα δώσει το κείμενό μου. Εμείς σας ε, ευχαριστώ. Ελπίζω πάντως με την απαραίτητη αυτή ανεξαρτησία θα γίνει καλύτερη αυτή η δουλειά. Ελπίζω λοιπόν να απασχολήσει αυτό το θέμα και το Συμβούλιο Ιδέα Απασχόληση Εξωτερικών Συμβούλων είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί η ανεξαρτησία τους δεν μπορεί να αξιολογηθεί από το Κοινοβούλιο. Επίσης έχουμε πει πως θα πρέπει να υπάρξει περιορισμός του διοικητικού βάρους, του άχθους. Συχνά σχετίζεται το Κοινοβούλιο με υπερβολική γραφειοκρατία και προτείνεται βεβαίως να μειωθούν αυτά κατά 30% αλλά ακούω και μηνύματα πως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτό οδηγεί στη μείωση των στάνταρτς από ε, των προδιαγραφών από πλευράς των επιχειρήσεων. Γι' αυτό πρέπει να το δει σφαιρικά αυτό το θέμα η Κομισιόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται εις βάρος ε, των ε, προδιαγραφών. Υπάρχει επίσης και ομάδα υψηλού επίπεδου υπό τον κύριο Στόιμπερ που βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπω πως επεκτάθηκε εντολή μέχρι το 2013 και οπωσδήποτε θα ενημερωθεί το Κοινοβούλιο για το πώς η ομάδα αυτή βλέπει τη μείωση των βαρών αυτών και τέλος να αναφέρω πως ε, η θέση ενισχύ της συνθήκης Λισαβόνας μας οδηγεί να δούμε πώς θα εμπαθυνθεί η επαφή με τα εθνικά κοινοβούλια και ελπίζω βεβαίως να μην περιοριστούμε εδώ πέρα μόνο στον έλεγχο της επικουρικότητας αλλά και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Τώρα οι πρωτοβουλίες πολιτών, θεωρώ πως εκατομμύρια πολιτών αναμένουν την στάση του Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζω πως το επεξεργάζεται αυτό Κομισιόν και ελπίζω να γίνει η πρώτη ανάγνωση ήδη φέτο και αναμένω τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε και τώρα τον λόγο θα έχει ο αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Σεύκοβιτ, έτσι ώστε να μα εξηγήσετε για τη θέση τη Επιτροπή επί του θέματο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την κυρία Γκέργκερ Ντεόντεμπερ για την άρεστη έκθεσή τη. Ευχαριστούμε και για όσα είπε καταρχήν με τα οποία και συμφωνεί η Επιτροπή διότι πάρα πολύ μας αρέσει το πόσο ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, η ευφύης αυτή νομοθεσία. Την Τρίτη θα πρέπει να σας πω ότι 59 ε, εκκρεμούσες προτάσεις της ε, αποσύρουμε που αφορούσαν κάποια προγράμματα. Δεν θα συνεχίσουμε την πρόθεση διότι βλέπουμε ότι πλέον ε, έχουν ξεπεραστεί γιατί έχει αλλάξει ο αρχικός ε, στόχος. Οπότε και έτσι προχωρούμε προς τι διαπραγματεύσει για την Συμφωνία Πλαίσιο. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι θα εγκρίνουμε αυτή την ανακοίνωση για την ευφυή νομοθεσία της 6ης ε, δεκάτου και επίσης ε, θα έχουμε και την ετήσια έκθεση ε, για την νομοπαρασκευαστική διαδικασία όπου θα δείξουμε και κάποια άλλα δευτερεύοντα ζητήματα οπότε και θα καλύψουμε τα όσα λέει στην έκθεσή τη, η κυρία Γκέριγκερ Ντιότεμπεργκ τώρα επειδή πιέζει ο χρόνος δεν θα τα πω όλα ξαντλητικά ξανικά κάποια συγκεκριμένα ζητήματα πρώτα πρώτα όλοι συμφωνούμε για την χρηματοπιστωτική κρίση και θεωρούμε ότι είναι αναγκαία, είναι σπουδαία η νομοθεσία ούτως ώστε να μπορεί να ευημερίσει μια κοινωνία και μια αγορά. Επίσης, όπως λέει η συγγήτρια, θα πρέπει να προσέξουμε για το πώς νομοθετούμε γιατί δεν θέλουμε να βαρύνουμε βιομηχανία ΜΜΕ με αχρίαστες διοικητικές ε, υποχρεώσεις ε, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και για τη μέλουσα αλλά και για την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένω, δουλεύουμε σκληρά, ούτω ώστε να συνεχίσουμε αυτέ τι τέσσερι βασικέ δραστηριότητε για την ευθύ νομοθεσία και θα συνεχίσουμε στην ίδια ρότα με τι μελέτε των επιπτώσεων να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε την νομοθεσία, να την απλουστεύσουμε και την υπάρχουσα ισχύουσα νομοθεσία, να μειώσουμε τις ε, υποχρεώσει τις διοικητικές για τις επιχειρήσεις και να κάτσουμε να αξιολογήσουμε ε, την νομοθεσία που ισχύει τώρα για να δούμε πόσο αποτελεσματική είναι. Επίσης πρέπει να σας πω ότι έχουμε κάποιες προστριβές και διαφωνίες. Θα σταθώ σε δύο θεματάκια. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά αυτό το σώμα, το ανεξάρτητο το οποίο λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις μέλη της επιπτώσεων της Κομισιόν γιατί τις κάνει η Κομισιόν τις μελέτες και λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο. Τελικά το Κοινοβούλιο ελέγχει την ποιότητα της νομοθεσίας. Επίσης, έχουμε τώρα ανταλλαγή απόψεων και ανταλλαγές επιστολών σε επίπεδο Προέδρων Κομισιών και Κοινοβουλίου για να εξετάσουμε το τι ισχύει σήμερα μετά την ε, αλλαγή λειτουργίας του Κοινοβουλίου. για το πώς θα διαμορφωθεί τώρα το σκηνικό, το θεσμικό ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικότερα λόγω των θεσμικών αλλαγών επίσης θέλουμε να υπάρχει καινοτομία που είναι καλό για επιχειρήσεις και τους πολίτες μέσω της πιο αποτελεσματικής νομοθεσίας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε. Επίτροπε Ταντέος Ζήφκα τώρα για την Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου στα πολωνικά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε κατά τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Χαίρομαι για το ότι και οι δικές μου παρατηρήσεις ελήφθαν υπόψη από την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Κοιτάξτε, στα πολλά αυτά χρόνια, πρώτα στην κοινότητα και τώρα στην Ένωση, καταλήξαμε στο ότι λειτουργεί η ευρωπαϊκή ρύθμιση όταν χρειάζεται να ρυθμίσουμε ένα θέμα σε 27 κράτη-μέλη. Βεβαίως, νέα νομοθεσία μπορεί να αποτελέσει και κάποιο είδους εμπόδιο, οπότε πρέπει να απλοποιούν τα πράγματα και να μην τα κάνουν πιο πολύπλοκα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους πολίτες να μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα νομικά κείμενα χωρίς αυτό να σημαίνει πώς θα πρέπει να μειώσουμε τυχόν προδιαγραφές. Αντιθέτως πρέπει να πάμε προς μια βελτίωση. Είναι πάρα πολλές αλλαγές μέσω της ε, συνθήκης της ε, Λισαβόνας που έχουν επίδραση στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου, οι πρωτοβουλίες ε, πολιτών, κατάργηση βαρών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα βοηθήσουν τους πολίτες και την ποιότητα της νομοθεσίας. Μεγαλύτερη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων θα οδηγήσει επίσης σε μεγαλύτερη ευθύνη έναντι των συμπολιτών μας. Το Κοινοβούλιο κέρδισε σε πραγματική επιρροή τη, στην νομοθεσία. Γι' αυτό πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τους βουλευτές και με τις ανεξάρτητες μελέτες επιπτώσεων και νομίζω εδώ πέρα σωστά έχει τονίσει την αποστολή της Κομισιόν η συγγήτρια. Πρέπει όμως να υπάρχει μια αναλογή βάση και για το κόστος και για τη μελλοντική εφαρμογή. Η καλή νομοθεσία είναι εγγύηση για την περαιτέρω εφαρμογή των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου στα κράτη-μέλη. Κάτι το οποίο βέβαια είναι δύσκολο. Ευχαριστούμε κύριε Σβίφκα. Και τώρα οι αγορητές ε, εκ μέρου των πολιτικών ομάδων και πρώτο, για δύο λεπτά για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κ. Μπαλτασάρη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η έκθεση της κυρία Γκέριγκερ υπογραμμίζει το βασικό πρόβλημα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την ανάγκη να υπάρξει μια απλή και διαφανής και κατανοητή νομοθεσία για όλου του πολίτε τη Ένωση. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τους στόχους τους οποίους ε, σημειώνει η συγγήτρια ο σεβασμός των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας η σημασία που δίδεται στις μελέτες των επιπτώσεων και ιδιαίτερα για αυτές θα ήθελα να πω ότι η Νομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εργάζεται ενεργά έτσι ώστε να πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει την ανάλυση και την ανεξαρτησία της ανάλυσης η οποία γίνεται κάθε φορά. Η ακαιρεότητα και η αντικειμενικότητα αυτών των μελετών θα βελτιώσει την ποιότητα των προτάσεων και θα επιταχύνει το χρόνο έγκρισης. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να μειώσουμε και το διοικητικό βάρος, σεβόμενοι βέβαια το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μειώσει κατά 25% μέχρι το 2012. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα 150 δις, δηλαδή ένα 0,5 αύξηση του ΑΕΠ. Φοβάμαι ότι η ανεπάρκεια των διαδικασιών των διοικητικών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο είναι υπεύθυνε. 72 σαν παράδειγμα νομικές πράξεις ε, επέβαλαν 470 υποχρεωτικές δημοσιεύσεις εφαρμοστικών διατάξεων. Όλα αυτά λοιπόν είναι απαραίτητα και σίγουρα απαιτούνται περισσότεροι έλεγχοι κατά την ε, πρώτη φάση της επεξεργασίας των νομικών ε, θέσεων και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι απαιτείται μεγαλύτερη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και αυτό θα βοηθήσει έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια νομοθετική δραστηριότητα πιο αποτελεσματική και πιο ε, θα έλεγα γειτονική στις πραγματικές ανάγκες του πολίτη. Ευχαριστούμε κύριε Βαλτασαριό, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το λόγο κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγγήτριά μας, η Λιδία Γκέριγκερ, υπέβαλε μια φιλόδοξη έκθεση. Εάν όλοι όσοι συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία τα τηρήσουν αυτά, έχουμε κερδίσει πάρα πολλά πράγματα και για την αξιοπιστία του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα πρέπει να βελτιωθεί το γενικότερο περιβάλλον, το ρυθμιστικό. Μιλάμε για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Δύο στοιχεία τη έκθεση είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η απλοποίηση του δικαίου δεν πρέπει να οδηγήσει στο ότι θα πέσουν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οπότε θα πρέπει να συνοδευτεί από μια άλλη πρωτοβουλία που θα λέγεται έξυπνη νομοθεσία. Κάθε νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να λαμβάνει ε, χώρα μετά από διαβούλευση των ενδιαφερομένων, ειδικά όταν έχει αντίκτυπο στην πολιτική απασχόλησης και την κοινωνική πολιτική επιπλέον θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα σοβαρό αξιολόγησης αντικτύπου. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα από το οποίο θα προκύπτει σαφώς πως η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία των μέτρων αυτών είναι εγγυημένη. Νομίζω πως στο παρελθόν είχαμε κάποιες άσχημες εμπειρίες. Σας σκεφτούμε εδώ πέρα την την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες και την αξιολόγηση που είχε κάνει τότε η Κομισιόν. Επίσης, η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει οριζόντιες ε, αξιολογήσεις αντικτύπου. Θεωρώ πως το σύστημα αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή, όπως αναφέρθηκε ήδη, να υπάρχει δηλαδή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για το, τις επιπτώσεις που έχει στην απασχόληση και τα κοινωνικά. Ευχαριστούμε. Για τους φιλελεύθερους τώρα. Για δύο λεπτά. Κυρία Τάιν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Τι εννοούμε καλύτερη νομοθεσία. Θέλουμε απλούστερη, πιο διάφανη και κατανοητή νομοθεσία για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαντικό είναι εδώ πέρα να γίνονται σεβαστές οι αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Δηλαδή θα ρυθμίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το οποίο δεν ρυθμίζεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σημαντικό κομμάτι της καλύτερης νομοθεσίας βεβαίως είναι ακριβώς το πώς θα επιδράσουν οι διατάξεις αυτές. Μόνο έτσι μπορούμε να περιορίσουμε τις τυχόν αρνητικές επιδράσεις. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πολύ καλή προετοιμασία από πλευράς Κομισιόν και είναι σημαντικό πως συναισθήθη με τα πίεση του Κοινοβουλίου ένα ανεξάρτητο συμβούλιο που θα κάνει αυτή την αξιολόγηση αντικτύπου, το οποίο όμως θα δίνει λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις επιχειρήσεις και τις αρχές και τους πολίτες. Η διατάξεις αυτές σημαίνουν κόστος, είτε σημαίνουν σήμανση προϊόντων, είτε οτιδήποτε άλλο. Και αν το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, καταργεί τον στόχο της πολιτικής. Θα πρέπει λοιπόν μέχρι το 2012 να μειωθεί η γραφειοκρατία κατά 25% και το διοικητικό κόστος. Αυτό λοιπόν σημαίνει πως θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά πρέπει εδώ πέρα να πούμε πως ένα τρίτο, ίσως και δύο τρίτα του διοικητικού βάρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτελέσμα αποφάσεων των κρατών μελών, τα οποία στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου επιτρέπουν πάρα πολλές άχρηστες και αχρίαστες διατάξεις. Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστεί η αχρίαστη γραφειοκρατία, θα πρέπει να ελέγξουμε την εφαρμογή του εθνικού δικαίου και ειδικά και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να ασκήσουν τη δυνατότητα και υποχρέωσή τους για να το κάνουν αυτό. Εμεί ευχαριστούμε και τώρα για του πρασίνου. Για ένα λεπτό. Η κυρία Λίχτενμπεργκερ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όταν θέλουν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα 27 διαφορετικά νομικά συστήματα, προφανώς θα υπάρχουν δυσκολίες. Εξού και η κριτική προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Η αντίδραση αυτή πρέπει να περιέχει κάποια βασικά σημεία όπως παραδείγματο χάρη εξιολογήσει αντικτύπου που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητος και θα λαμβάνει υπόψη όλους τους ενδιαφερόμενους, όχι μόνο τη βιομηχανία και τα λόμπι. Αυτό είναι σημαντικό για εμένα. Το άλλο είναι η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Πάρα πολλέ δυσκολίες προκύπτουν ακριβώς στη φάση της εφαρμογής ή μη εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς εδώ όταν μιλάμε για την εφαρμογή να επιφέρουμε βελτιώσεις και να βασιστούμε σε πολίτες οι οποίοι θα αντιδρούν με τρόπο αποτελεσματικό και κοινοτόμο. Νομίζω πως οι αντιδράσεις των πολιτών έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Για συντηρητικού μεταρρυθμιστέ, έχει το λόγο για δύο λεπτά ο κύριο Καρίν. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια ε, για την εκθεσή τη για το ότι μα εκάλυψε σε πολλά που θέλαμε, γιατί νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση η καλή βελτίωση της νομοθεσίας για το μέλλον όλων των κρατών και πάρα πολλά από τα νομοθετήματα που κάνουμε ε, βέβαια δεν πιάνουν τόπο και πρώτα πρώτα διότι έχουμε ένα σωρό κανονισμούς που δεν χρειάζονται και συνεχίζουν όμως να ισχύουν οπότε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο διοικητικό βάρο ε, και βαρύνει τη ΜΜΕ που αποτελεί τη ποδηλική στήλη τη ε, οικονομία μα και πάρα πολύ θετικό το ότι αυτό το αναγνωρίζει η Κομισιόν. Κάτι άλλο, είπα ότι έχουμε κάποιε τρελέ πρωτοβουλίε τη Κομισιόν που τι έρχονται από ακυρού καιρών και με αυτόν τον τρόπο το μόνο το οποίο καταφέρνουμε είναι να μην επιτελούμε το έργο που πραγματικά χρειάζεται. Τώρα, αν κάνουμε τώρα κάποια βήματα πέρα από τη στιγμή της Λισαβόνας ε, θα πρέπει να μην ξεχνούμε κάποια ζητήματα τα οποία επισημάνθηκαν από τους συναδέλφους πρώτα-πρώτα ε, είμαι για την επικουρικότητα και για την αναλογικότητα ε, μόνιμος εισηγητής και πρέπει να σας πω ότι τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία όμως χρειάζεται να υπάρχει και η αντίστοιχη ερμηνεία και τέτοιου είδου υποστήριξη. Αλλιώ δεν μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Τώρα, όσον αφορά τι μελέτε των επιπτώσεων, χαιρετίζουμε τι εξελίξει και ότι χρειάζονται διαβουλεύσει με όλου του ενδιαφερομένου. Χρειάζεται συμμόρφωση προ την αρχή τη υπογερικότητα. Αυτό κάθε φορά να εξετάζεται και πάρα πολύ σωστό είναι αυτό που λέει η έκθεση για θα πρέπει να δοθεί κάποιο ορισμό τη έννοια τη ευφυή νομοθεσία και θα πρέπει να υπάρχει η μελέτη των επιπτώσεων ευθύς εξ αρχής και να μπορεί το Κοινοβούλιο από την αρχή να, να συνοηθεί πριν γίνει οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση με την Κομισιόν. Η πολιτική μας ομάδα επίσης θεωρεί ότι είναι θετικό το ότι προχωρούμε με αφετηρία το ότι οι ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να σεβαστούν αναλογικότητα και επικουρικότητα και ότι θα πρέπει κάθε ε, νομοθέτημα να ε, λαμβάνει αυτού το υπόψη και το ότι θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε μια μελέτη επιπτώσεων που θα πρέπει να γίνεται με τρόπο αμερόληπτο και θα πρέπει ε, να υπάρξει ενόηση κοινοβουλευτικών επιτροπών και κομισιών και έτσι να προσπαθούμε να πλησιάσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον Ευρωπαίο πολίτη. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε και τώρα για την Ευρώπη της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Μέσερ Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αναφέρθηκαν πάρα πολλά σημαντικά σημεία και ιδιαίτερα βεβαίως αυτά που αφορούν αναλογικότητα και επικουρικότητα. Δυστυχώς οι προθέσεις ε, στην ε, συνθήκη της Λισαβόνας με στιγμής δεν έχουν μεταφραστεί σε κάτι απτό. Κάτι το οποίο είναι λυπηρό εάν δούμε ε, το πώς υπάρχει αυτή η αρμοδιότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων η οποία όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί και βλέπουμε πως ε, κάποια κοινοβούλια θέλουν εάν θέλουν κάποια κοινοβουλία να σταματήσουν την νομοθεσία γιατί δεν είναι αναλογική, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να το κάνουν και όχι να έχουν αυτές τις κίτρινες κάρτες. Αυτό είναι αστείο και είναι λυπηρό να ηρωνευόμαστε έτσι την κυριαρχία των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Τώρα, ας ε, επικεντρωθούμε στις στοιχείες που έχουμε μπροστά μας. Ελπίζω η Κομισιόν να καταλήξει σε μια κατάσταση στην οποία θα γίνονται σεβαστά τα κράτη-μέλη και δεν θα ενημερώνονται απλώς για το τι ε, θεωρούν ε, τα κράτη-μέλη για την νομοθεσία. Μην γεγραμμένη τώρα στο Γιάννοφ. μιση λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προηγούμενους συναδέλφους ιδιαίτερα σχετικά με τις δυνατότητες που θα έχουν πλέον τα κοινοβούλια των κρατών μελών που αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες και που μπορούν να παρέμβουν σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας όταν κρίνουν τα κοινοβούλια αυτά ότι υπάρχει μια μη ικανοποιητική κατάσταση. Αυτό είναι ένα θετικό κομμάτι της συνθήκης της Λισαβόνας. Διαρωτώ όμως αν δεν ήταν παρά ένα λαϊκιστικό μέτρο μόνο και μόνο για να προκαλέσει περισσότερη υποστήριξη θα έλεγα. Γιατί αν πράγματι δίδονται νέες αρμοδιότητες στα κοινοβούλια των κρατών μελών τότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δημιουργηθεί μια διαδικασία, να καθοριστεί μια μέθοδος σύμφωνα με την οποία τα κοινοβούλια των κρατών μελών μπορούν να συνεργάζονται, μπορούν να συντονίζονται και να εργάζονται από κοινού γιατί αυτή η απέτηση που υπάρχει τα δύο τρίτα των ε, κοινοβουλίων των κρατών μελών ε, που θα πρέπει να συμφωνούν για να προχωρήσει μια τέτοια διαβούλευση είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Απαιτείται λοιπόν μια συνολική διαδικασία για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προς την Βελγική Προεδρία η οποία θα φιλοξενήσει τη συνάντηση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Μας είπε. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται, προκύπτει και πάλι και, κάθε χρόνο κουβεντιάζουμε τα ίδια και τα ίδια και θυμάμαι ότι είχε καταβληθεί μια προσπάθεια από την Μόνικα Φρασόνια, τον Μεδίνα Ορτέγα σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές θητείες. Όμως, συγχαρητήρια για την παρούσα έκθεση από την οποία θα πρέπει να προσέξουμε όχι μόνο αυτά τα οποία αναφέρει, όχι μόνο τους στόχους, αλλά και το πνεύμα αυτής της έκθεσης. Αυτό θα πρέπει να διαπνέει κάθε πράξη όλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς, για άλλη μια φορά, θα επαναλάβουμε τα ίδια κουραστικά για το τι γίνεται, για το ποια είναι τα δεινά που μας ταλαιπωρούν, για το τι λάθη κάνουμε. Επομένω, γι' αυτό σα λέω ότι θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα οποία είπε ο κύριο Επίτροπο, που δεν είναι μόνο θέμα βολονταρισμού. Είναι θέμα αξιοπιστία, κύριε Επίτροπε. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που καταβλήθηκε με αυτή την έκθεση μπορεί να πιάσει τόπο για να πετύχουμε ε, το στόχο του 25% και όλα τα άλλα τα οποία τάση ο στόχο αυτή η έκθεση και για το πνεύμα τη. Πρέπει να προσέξουμε. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω στην έδρα του, στο έδρανό τον κύριο Σιμάνσκι. Αλλού είναι, όχι δεν είναι αλλού. Επομένω τώρα για 1,5 λεπτό έχει το λόγο ο κύριο Έρενχάουζερ. Θα ήθελα να πω κάποια λόγια για την αρχή της επικουρικότητας. Βεβαίως πρέπει η πολιτική επί της αρχής να βρίσκει, να λαμβάνει χώρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και μόνο τότε μπορεί να ελέγξει την ε, πολιτική ο πολίτης και μόνο έτσι μπορεί να ασκήσει και την άμεση δημοκρατία. Και αυτό ακριβώς είναι το νόημα της αρχής της επικουρικότητας. Εξού και η αιτιολόγηση που απαιτείται. Πρέπει δηλαδή με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια να επιχειρηματολογήσουμε και να πούμε γιατί η πολιτική πρέπει να ασκηθεί στο ευρωπαϊκό και όχι στο τοπικό επίπεδο. Όμως η κατάσταση έχει ως εξή και αυτό θέλω να αναφέρω. Αυτή η αιτιολόγηση, η ανάγκη αιτιολόγησης συχνά περιφρονείται. Βρίσκουμε εκεί πέρα αιτιολογήσεις ε, που λέγεται πως η πολιτική αυτή θα ασκηθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν επιχειρήματα δηλαδή γιατί να ασκηθεί γιατί ασκείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για το δικαίωμα ελέγχου της επικουρικότητας ε, που έδωσε η συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν επαρκεί αυτό. Δεν έχουν αρκετή ισχύ τα εθνικά κοινοβούλια και το δικαίωμα αυτό είναι μόνο στα χαρτιά. Και απαιτώ Άρα από την Κομισιόν ε, να δει πολύ εντονότερα την αιτιολόγηση αυτή της επικουρικότητας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω στο έδρανο της ούτε την κυρία Τσίλντες. Άρα θα δώσουμε το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Κοζούσνικ. Πολωνικά. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για την υψηλή ποιότητα η έκθεση. Για να σας πω δύο λόγια επ' αυτού. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάποια σημαντικά βήματα τόσο να βελτιωθεί η νομοθεσία. Παρ' όλα αυτά, δεν είμαστε τόσο ευχαριστημένοι όσο θα μπορούσαμε να είμαστε, γιατί πολλές φορές εδώ υπάρχει διχογνωμία σε σχέση με το Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Υπάρχει αυτή η ομάδα εργασία, ούτω ώστε να περισταλεί η γραφειοκρατία. Έχουμε το έργο του κυρίου Στόιμπερ επ' αυτού και θα πρέπει να σταθούμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο αυτή τη έκθεση. Εκεί που αναφέρει η γήτρια ότι θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμό των υπαλλήλων που ασχολούνται με την με, τη, με τις, με τις ε, μελέτες των επιπτώσεων θα μπορούσαμε εμείς να βοηθήσουμε την κατάσταση με το να κάνουμε και εμείς ε, μελέτη επιπτώσεων και θα βοηθούσαμε το αρμόδιο όργανο της Κομισιόν έτσι θα είχαμε περιστήλει και τις σχετικές δαπάνες τα θεσμικά οργάνα για τα δύο Ευχαριστώ συνάδελφε λέει ο Πρόεδρος Ούτε ο κ. Σιμάνσκι, ούτε η κυρία είναι στο έδρανό του από ό,τι βλέπω και επομένω τώρα πάμε ε, στο, στο, στο γύρο των παρεμβάσεων που λέγεται Catch the Eye. Όπως ξέρετε θα έχετε μόνο ένα λεπτό για να το υπερβείτε πρόκειται να σα αφαιρέσω το μικρόφωνο. Ο κύριο Μέσαρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν είπατε σωστά το όνομά μου. Εν πάση περιπτώσει να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας μπήκαμε σε μια νέα εποχή και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα κοινοβούλια. Ο ρόλος μας είναι πολύ μεγαλύτερος και έχουν αυξηθεί και οι ευθύνε μας και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε επιθανή δυνατότητα έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ομοθετική διαδικασία και παραγωγή. Υπάρχουν δύο σημεία τα οποία έχουν σχέση με τις μικρομεσαίες και έχουν πολύ μεγάλο βάρος για το κατά πόσον θα τις διαβουλευόμεθα. Θα πρέπει να υπάρχουν αιτίε για την συγκεκριμένη νομοθετική δραστηριότητα, θα πρέπει να υπάρχει απλούστευση της υπάρχουσας δραστηριότητας και θα πρέπει να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει επίσης να διαβουλευόμεθα και με τα κοινοβούλια των κρατών μελών. Μέχρι τώρα η στάση μας επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στην νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, καλύτερη νομοθεσία. Αλλά η μέθοδος που έχουμε δεν αποδίδει. Γιατί τι γίνεται με τα περιφερειακά ή τα κρατικά κοινοβούλια. Από τότε που άρχισε να ισχύει η καινούργια έχει να η καινουργια συνθηκη ανατέθηκαν 26 πρωτοβουλίες στα κοινοβούλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα 27 αυτές πρωτοβουλίες ε, αφού 27 κράτη πήραμε 52 ε, από τις 72 δυνατές απαντήσεις περίπου 7% την ανταπόκριση και από αυτά τα 52 ε, τα 10 ε, ήταν από την Αυστρία ένα από την Τσεχία, ένα από την Ισπανία ένα από τη Γαλλία ε, τρία, τρεις από το τελικό κοινοβούλιο ε, από την Πολωνία και από την Πορτογαλία και από τις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν μας δίνει τίποτα στοιχεία για τη συμμετοχή των περιφερειακών κοινοβουλίων όσον αφορά αυτά τα νομοθετήματα. Αυτά όλα τα προβλήψει της Λισαβόνα. Ευχαριστούμε κύριε Βιλβάλη. Ο πρόεδρος που της αφαίρει το λόγο και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ρούμπιχ. Paldies, priekšsēdētāji. Es visumā ar gandarību. Συνολικά η δομένη κατάσταση νομίζω ότι είναι θετική και συμφωνώ με την έκθεση. Κοινοβούλιο αλλά και γενικότερα Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να ισχύσουν τα όσα θέλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτό αυτή όμω θα πρέπει το ίδιο να γίνεται αυτό που ζητούμε δηλαδή από του απέξω γίνεται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θέλω να παρατηρήσω ότι πολλέ φορέ δεν υπάρχει απαραίτητη εποπτεία. Έχουμε κάποια νομοθετήματα τα οποία δεν εφαρμόζονται σε αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να ξεκαθαρίσουμε το εξή το οποίο συνέβη στις 2 ε, Οκτωβρίου η Λετωνία πρόκειται να κάνει κοινοβουλευτικές εκλογές, η χώρα μου. Ή αυτέ αυτές τις εκλογές που θα διεξαγάγουμε και αφαιρείται ο λόγος από τον ε, πρόεδρο που ξεπεράσετε το χρονικό όριο και το λόγο κυρίως Πάσκα.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 ďalšou dôležitou úlohou potom ešte bude zabezpečiť aj vytvorenie siete kvalitných akreditovaných inštitúcií špecializovanej prípravy odborníkov mr president the legislative process as it η νομοθετική διαδικασία όπως λαμβάνει η χώρα εδώ πέρα φαίνεται πως έχει στόχο μέλη και τους βουλευτές να ασκούν οποιαδήποτε κρίση. Οι τροπολογίες ε, υπάγονται σε μεγαλύτερες ομάδες ε, τροπολογιών και βεβαίως όσοι ακολουθούν τις οδηγίες του κόμματός τους ε, δεν χρειάζεται να απασχολούν πολύ το μυαλό τους, αλλά οι ανεξάρτητοι βουλευτές ή μέλη μικρών κομμάτων που σκέφτονται και όλας πριν ψηφίσουν πρέπει να σκεφτούν τι θα κάνουν. Θα πάνε σε μια συζήτηση και θα λάβουν απόφαση ο βοηθός τους ή θα ασχοληθούν με την ομοθεσία για να λάβουν απόφαση. Ε, δεν γίνεται έτσι δημοκρατία. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Ε, προβλέπουν οι διαδικασίες ότι πέντε λαμβάνουν το λόγο για αυτή τη διαδικασία, αλλά κάτι εξαίρεση θα δουν το λόγο σε άλλους δύο. Πρώτα-πρώτα στην κυρία Κολάρσκα. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω την εισηγήτρια για την έκθεση αυτή. Πράγματι ε, έχει αντιληφθεί την ανάγκη να δημιουργηθεί σωστό δίκαιο. Βεβαίως ε, εμείς κάνουμε εκθέσεις, δηλώσεις με μία γλώσσα η οποία είναι τόσο δύσκολη και πολύπλοκη ώστε απλός κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα πάρα πολλά έγγραφα που παράγονται εδώ πέρα ε, πολύ απλά δεν είναι ευανάγνωστα και η γλώσσα είναι αποκλειστικά νομική και τα ψηφίσματα που συντάσσουμε επίσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα το ίδιο με την ίδια μορφή οπότε θα πρέπει το κοινοβούλιο να ακολουθήσει αυτό το οποίο κάνει και η Κομισιόν μία καμπάνια για να γράφουμε κατανοητά. Έτσι πρέπει να παράγουμε τα έγγραφα για να μπορούν να διαβάζονται. Και θα ολοκληρώσουμε αυτή τη φάση της συζήτησης με την παρέμβαση της κυρίας Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, Ήμουν στο γραφείο μου και παρακολούθησα από εκεί πολύ προσεκτικά τη συζήτηση και οπότε πρέπει να ευχαριστήσω την κυρία Γκέριγκερ αλλά και, και εσά κύριε Επίτροπε για τα όσα είπατε. Είναι νομίζω πάρα πολύ ευχαριστώ το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συνεκρότησε αυτήν την ομάδα υψηλού επίπεδου που θα παρέχει τις συμβουλές της ε, σε σχέση με την, την μείωση της ε, γραφειοκρατίας. Βέβαια κάθε χώρα έχει τη δική της κουλτούρα και παράδοση αλλά ο, πάρα πολύ σημαντικός ε, πολιτικός στόιμπερ ο οποίος τέθη επικεφαλής αυτής της ομάδας ε, εγγυάται ε, την επιτυχία γιατί είναι κάτι πάρα πολύ επιθυμητό η μείωση της γραφειοκρατίας. Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε. Και τώρα θα λάβει το λόγο ο αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς για να απαντήσει στα όσα είπαν οι ομιλητέ μα. Έχετε το λόγο κύριε Πίτροπο. Uh, Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να δώσω όσο περισσότερες απαντήσεις μπορώ μέσα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας που είναι περιορισμένος. Να ευχαριστήσω τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δείχνουν ότι η εξυπνότερη και απλούστερη νομοθεσία είναι κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο και θα καλύψει τις ανάγκες των κρατών μελών. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια γιατί πράγματι συμφωνούμε για τα θέματα των, με τα θέματα τα οποία υπογραμμίζει και προχρήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως οι μελέτες επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να βελτιωθούν, η ποιότητά τους θα πρέπει να βελτιωθεί, η αντικειμενικότητά τους είναι απαραίτητο στάδιο για την απλούστευση εκ των υστέρων της νομοθεσίας. Αυτό που έχει σημασία και υπογραμμίζεται στην έκθεση είναι ότι υπάρχει ανάγκη να μελετήσουμε τις συνέπειες των τροπολογιών. Ο νομοθέτης προτείνει μεν, αλλά κάποιες τροπολογίες οι οποίες μπορεί να γίνουν δεκτές σχετικά βιαστικά μπορεί είτε να βελτιώσουν την νομοθεσία είτε όμως και να την περιπλέξουν. Θα συμφωνήσω επίσης με αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι απαιτούνται ανεξάρτητες ε, μορφές ε, αξιολόγησης. Αυτό κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε και με τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες έτσι ώστε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και άνω του 30% των προτάσεων που γίνονται στις υπηρεσίες από την ε, υπηρεσία που ασχολείται με τις μελέτες επιπτώσεων απορρίπτονται. Για τις μικρομεσαίες έχουν συζητηθεί πολλές φορές τα προβλήματά τους για το πώς μπορούμε να μειώσουμε το βάρος ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. μέχρι το τέλος του 2012 θα πρέπει να μειώσουμε το βάρος αυτό κατά 25%. Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια πάντως, ε, να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που είναι υπέρ αυτής της εξυπνότερης και απλούστερης διαδικασίας. Κύριε Σεύκοβιτς. Δεν υπάρχει περιορισμός χρόνου για σας. Εσείς αυτό περιοριστήκατε. Ίσως δεν έπρεπε να σας το πω γιατί είναι κακό προηγούμενο, αλλά καλό είναι να πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν έχει χρόνο έτσι ώστε να αυτό ε, λογοκρίνεται σε εισαγωγικά. Ευχαριστώ κύριε Σεύκοβιτς. Το λόγο έχει η κυρία Γκέριγκερ Ντέντενμπεργκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους ε, και σα κύριε Επίτροπε για αυτή την ε, επικοδομητική συζήτηση. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το ότι είχα την ευκαιρία ειδικά φέτος να προετοιμάσω αυτή την έκθεση για την καλύτερη νομοθεσία. Την πρώτη δηλαδή χρονιά μετά την ε, θέση ενισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και την υποβολή της έκθεσης για το 2020. Βάρα, μίλησα με πολλούς ενδιαφερομένους και στον κόσμο της βιομηχανίας, των συνδικάτων, των εργαζομένων και των κλαδικών οργανώσεων τους όπως η ETUC. Ομόφωνα στην Επιτροπή μας ε, υιοθετήσαμε την έκθεση αυτή και βρήκαμε ένα καλό συμβασμό που ικανοποίησε τις προσδοκίες όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ λοιπόν την πολύ καλή αυτή η διακομματική συνεργασία κατά το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Ελπίζω λοιπόν να μπορούμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα και σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Και με αυτή την παρέμβαση ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψήφιση της εκθέσεως πρόκειται να γίνει το μεσημέρι με